πρέπει να συμμετέχουν μαζί με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τοποθετήσεις, όσον αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά αυτά θέματα. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας αυτά. Και τώρα θα σας δώσω γραπτός απάντηση σε αυτό που μου είπατε. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε στην έκθεση και το λόγο έχει συνάδελφ, είναι τη συναδέλφου μας της κυρίας Άννης ε, Ποδηματά και έχετε το λόγο κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όδης συζητητές, τη Γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και τους αρμοδίους των πολιτικών ομάδων για την ε, επικοδομητική συμβολή τους στις συζητήσεις και τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. η έκθεση πρωτοβουλίας του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης δεν θα μπορούσε να έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή γιατί η κρίση που θέτει σε δοκιμασία όπως γνωρίζουμε όλοι ιδιαίτερα σήμερα τη ζώνη του ευρώ έχει οδηγήσει σε σημαντική συρρήκνωση των δημόσιων πόρων σε εκτεταμένα προγράμματα λιτότητας και δημοσιονομικής εξυγίανσης από την πλειοψηφία των κρατών μελών και παράλληλα δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στον ίδιο τον κοινοτικό προπολογισμό, και αυτό το ζήσαμε πολύ πρόσφατα στη συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. προκύπτει ένα βασικό και κοινά αποδεκτό συμπέρασμα από την περιγραφή αυτής της κατάστασης οι ευρωπαίοι πολίτες είναι αυτοί που σηκώνουν το μεγάλο βάρος της κρίσης με τη συρρήκνωση των εισοδημάτων τους με την ανεργία με την ανασφάλεια που διέπει τις εργατικές τους σχέσεις και με την συρρήκνωση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. το δεύτερο βασικό και κοινά αποδεκτό συμπέρασμα που προκύπτει από την κατάσταση αυτή είναι ότι η ένωση και τα κράτη μέλη χρειάζονται επιγόντως νέους πόρους που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάκαμψη και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας αυτή τη φορά με τρόπο ισορροπημένο που θα περιορίζει τις ανισότητες και τις αποκλίσεις γιατί μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020 και μόνο έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά εύρυθμη και ισχυρή εσωτερική αγορά προς όφελος των πολιτών της. χρειαζόμαστε λοιπόν νέους πόρους και συμφωνούμε όπως ρητά αποτυπώνεται στην έκθεση και διαβάζω τη σχετική παράγραφο ότι η περαιτέρω αύξηση του ύψους και του εύρους των σημερινών φορολογικών εργαλείων όπως και οι περαιτέρω περικοπές των δημοσίων δαπανών δεν αποτελούν ούτε επαρκή ούτε βιώσιμη λύση για να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο επίπεδο τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης μπορούν να παίξουν ένα ρόλο κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών γιατί μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων σημαντικών εσόδων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. δεν είναι όμως μόνο αυτό ε, συνάδελφοι ε, το όφελος των καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης. καινοτομία στη χρηματοδότηση δεν σημαίνει απλά και μόνο ανέβρεση νέων πόρων εξίσου σημαντικό είναι να ανοίξουμε το δρόμο για μια σταδιακή αλλαγή του σημερινού φορολογικού μοντέλου όπου το κύριο βάρος της φορολόγησης και γενικότερα της χρηματοδότησης της οικονομίας πέφτει παραδοσιακά σε τομείς όπως η εργασία οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικές επενδύσεις. η σημαντική προστιθέμενη αξία των καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων το διπλό όφελος όπως λέμε είναι ότι εκτός από έσοδα μπορούν να έχουν και έναν ισχυρό ρυθμιστικό ρόλο να αποθαρρύνουν πρακτικές και συμπεριφορές επιβλαβείς είτε μιλάμε για το χρηματοπιστωτικό τομέα είτε μιλάμε για το περιβάλλον και την προστασία του. η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα τα ευρωομόλογα και τα ευρωπαϊκά επενδυτικά ομόλογα το φόρο άνθρακα και τη χρηματοδότηση για αναπτυξιακούς στόχους σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ξεκινάμε πάλι από μια βασική και κοινά αποδεκτή παραδοχή ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας αν και έχει τη βασική ευθύνη για την κρίση αν και δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί παρά την κρίση υπερκέρδη υποφορολογείται καθώς εξαιρείται σχεδόν καθολικά από το φόρο προστιθέμενης αξίας. μια δεύτερη επίσης κοινά αποδεκτή παραδοχή που προκύπτει απλά και μόνο αν δει κανεί τα νούμερα τα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε και γιγαντώθηκε ο όγκο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία είναι η μεγάλη και συνεχώς διευρυνόμενη απόκλησή του από το βασικό του ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. οι δύο αυτές παραδοχές είναι ευρέως αποδεκτές από το κοινοβούλιο αλλά και από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέσω της πρόσφατης ανακοίνωσής της για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια καταφανή αδικία που πρέπει να αποκατασταθεί. You είχατε δύο τμήματα όσον αφορά το χρόνο σας. Αν θέλετε να μιλήσετε κι άλλο ένα λεπτό, καλώς αλλά στο τέλος δεν θα έχετε χρόνο να δευτερολογήσετε. Thought... Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ποδηματά, έλεγα ότι είχα πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά στην αρχή θεωρούσα ότι είχα. Ε, έχουμε να κάνουμε με μια καταφανή αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί, στέλνοντας και ένα ισχυρό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες ότι όντως έχουμε αντλήσει διδάγματα από την κρίση, ότι επιδιώκουμε το δικαιότερο επιμερισμό των βαρών και ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να επανέλθει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στο βασικό του ρόλο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. υπάρχει μια ευρεία συνένεση ότι το πλέον κατάλληλο φορολογικό εργαλείο για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί με αυτό το φόρο το φορολογικό βάρος είναι συνάρτηση της ποσότητας της συχνότητας και τελικά της ποιότητας δηλαδή της προστιθέμενης αξίας της ίδιας της συναλλαγής γιατί όπως σημειώνουμε όλοι μαζί με συμφωνία στην παράγραφο 13 ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των πιο επιβλαβών πρακτικών στις συναλλαγές όπως είναι οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας και να περιορίσει την κερδοσκοπία είναι προφανέ ότι η πρώτη επιλογή όλων μας είναι να θεσπιστεί ο φόρος αυτό σε παγκόσμια κλίμακα όμως είναι εξίσου προφανέ ότι παρά τις αρχικά φιλόδοξες δηλώσει αντί να ενισχύονται οι πιθανότητε για μια παγκόσμια συμφωνία συνεχώς περιορίζονται. το ερώτημα λοιπόν αγαπητέ συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι είναι τι κάνουμε εμεί στην ευρώπη. κρυβόμαστε πίσω από την έλλειψη παγκόσμια συμφωνία είναι αυτό αρκετό και κυρίως είναι πιστικό για τους πολίτες μας που επομίζονται το βάρος τη της Ακόμα και αν αυτό δεν είναι, εύκολο να συμβεί, γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου σε αυτό το θέμα, ακόμα και αν υπάρχουν... Mr. President, I had seven minutes and uh, Κύριε Πρόεδρε, είχα, είχα 7 λεπτά. Έχω ακόμα 30 ε, δευτερόλεπτα. Τέσσερα συν δύο μου έχουν σημειώσει εμένα εδώ πέρα. Πέντε συν δύο, λέει η κυρία Ποδηματά. Okay, Συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να, για να ολοκληρώσω, ότι ακόμα κι αν δεν είναι εύκολο να προχωρήσουμε άμεσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο στη θέσπιση φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί δεν είναι εύκολο να υπάρξει ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ως το μόνο ευρωπαϊκό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους ευρωπαίους πολίτες έχει υποχρέωση να στείλει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα προς την κατεύθυνση αυτή. είναι δική μας ευθύνη να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα δεν είναι ευθύνη της ευρωπαϊκής επιτροπής. ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Επιτροπές Οικονομικών και Ανάπτυξης και ειδικά την κυρία Άννη Ποδηματά για την έκθεσή της για την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχα ήδη την ευκαιρία να συζητήσω αρκετές φορές μαζί σας το πώς θα κάνουμε τις τράπεζες να πληρώσουν το κόστος της κρίσης. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν προετοιμάζει μια αξιολόγηση αντικτύπου εις βάθος για τα μέσα φορολογίας του χρηματοπιστωτικού τομέα με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2011. Έτσι θα μπορέσει η Κομισιόν να υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για δράσεις πολιτικής. Επίσης εξετάζουμε το σωρευτικό αποτέλεσμα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των νέων φόρων και τελών και θα παρουσιάσουμε και εισφορών και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αργότερα φέτος. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να περιμένετε αυτά τα αποτελέσματα πριν λάβετε οποιαδήποτε θέση για την εισαγωγή φόρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τη φορολογία του άνθρακα, συμφωνώ πως το τωρινό μοντέλο φορολόγησης ε, δεν εφαρμόζει πλήρως στην αρχή ορυπένων πληρώνει. Καλωσορίζω τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση του στήματος εμπορίας εκπομπών καθώς και για την συνολική αναθεώρηση της οδηγίας φορολόγησης ενέργειας έτσι ώστε να γίνει το περιεχόμενο της ενέργειας ε, το βασικό κριτήριο φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων. Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας αυτής ε, έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2011 επίσης. Άκουσα τις ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους διαρροής άνθρακα. Εμείς είμαστε υπέρ ε, μεταβατικών δωρεάν παροχών αδείας και πρόσβαση σε διεθνείς άδειες ε, υπό το σύστημα εμπορία. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούμε να παρακολουθούμε του τωρινού και μελλοντικού κινδύνου διαρροή άνθρακας και είμαι, άνθρακα και είμαι επιβεβισμένος πω μια τέτοια δωρεάν παρχή αδειών υπό το σύστημα αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση τη οδηγία. Τέλο, όσον αφορά τα ευρωομόλογα, η Κομισιόν αναγνωρίζει πώ ανάλογα με τι ακριβείς λεπτομερείς η κοινή έκδοση ευρωομολόγων θα μπορούσε να ευνοήσει την αποτελεσματικότητα των ε, αγορών ομολόγων και τη στήριξη του ευρώ ως ε, διεθνούς νομίσματος. Όμως πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ανάλυση και συζήτηση σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο συγκεκριμένα το τι σημαίνει αυτό για το ηθικό ρίσκο των κρατών, τον ηθικό κίνδυνο των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε κύριος Μαριάν Μαρινέσκο από την Επιτροπή Έρευνας και ε, Βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επίτευξη των στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, κλιματικέ αλλαγέ, όλα αυτά απαιτούν σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση, ιδίω για την καινοτομία και την έρευνα, αλλά και για νέου τρόπου ώστε να εξεύρουμε την ε, χρηματοδότηση που απαιτείται. Μιλήσατε για τη σκοπιμότητα εισαγωγή ενός φόρου άνθρακα που θα μοιάζει με το ΦΠΑ και θα επιβάλλεται σε κάθε προϊόν που κινείται στην αγορά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του φόρου αυτού μεταξύ των συνόρων και θα πρέπει να βοηθήσουμε βέβαια και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα τα διαρθωτικά ταμεία, καθώς και τους ε, πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ εθνικών, ευρωπαϊκών ταμείων και άλλων μοχλών στήριξης που θα δίνουν και κίνητρα για ενεργειακή απόδοση και καινοτομία. Οι ε, παρκείς επενδύσεις επίσης για τον ενεργειακό εφοδιασμό, την ενεργειακή απόδοση θα μειώσουν ε, την εξάρτηση, την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης και θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το συντομότερο δυνατό λοιπόν θα πρέπει να εκπονηθεί αυτή η μελέτη επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε και ποιο οικονομικό όφελος θα υπάρξει από τη μείωση των κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διαστρεβλούν σοβαρά την αγορά. Θα πρέπει η μελέτη αυτή επίση να αναλύσει κατά πόσον ο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι και ένα ίδιο πόρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you ευχαριστώ πολύ εκ μέρους του ΕΛΚ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Ζαν ε, Πολ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς δύο παρατηρήσεις ε, για τη μορφή. Η συγγήτριά μας επικρότησε το έργο όλων αυτών οι οποίοι συνεισέφεραν ε, στην έκθεση. Και πράγματι έγινε σημαντική δουλειά συντονισμού και η κυρία Χούπνερ που ήταν σκιώδη συγχύτρια από την ε, δική μας την Επιτροπή τα κατάφερε πολύ καλά. Όμως η σοσιαλιστική ομάδα έμαθα ότι έχει καταθέσει ένα αλλακτικό ψήφισμα. Σημαίνει αυτό ότι θα ψηφίσουμε καταρχάς ένα κείμενο το οποίο, για το οποίο δεν έγινε καμία διαβούλευση. Δεύτερη παρατήρηση πολιτικού ε, χαρακτήρα και δεν είναι στο χαρακτήρα μου ε, νομίζω ότι υπάρχει μια τεχνητή αντίθεση και αντιπαράθεση, ιδίω ό,τι αφορά το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Η δική μα ομάδα έχει σαφή θέση. Είμαστε υπέρ ενό νέου φόρου, ε, τέτοιου φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε υπέρ να πειραματιστεί με το φόρο αυτό η Ευρώπη, αν αυτό δεν καταστηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να λαμβάνουμε τέτοιε αποφάσει χωρί να έχει προηγηθεί μια σοβαρή μελέτη επιπτώσεων, η οποία θα επιτρέψει να διαπιστώσουμε κατά πόσο η ανταγωνιστικότητα των χρηματιστηρίων ε, υποστεί κάποιε αλλιώσει. Θέλω να πω τέλο, κύριε Επιτρόπε, τη θέση του ΕΛΚ δεν είναι μια θέση για να κερδίσουμε χρόνο, δεν είναι θέση αναμονής. Εμείς ζητούμε επιμόνως και με τα την μελέτη αυτή επιπτώσεων. Το έχουμε συζητήσει και ζητήσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο και θέλουμε να γίνει ε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η μελέτη αυτή για να μας διαφωτίσει. Έχουμε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 Εδώ και μήνες έχετε την εντολή από το Κοινοβούλιο να εξετάσετε με ποιον τρόπο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε για έναν φόρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δεν το κάνατε μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε για τη θέση σας, μας το έχετε πει και πολλές φορές γραπτός, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο θα θέλατε είναι να φορολογήσουμε τις μικρές τράπεζες που ακόμα έχουν υποκαταστήματα, που ασχολούνται με πελάτες, με επιχειρήσεις που δίνουν ακόμα δάνεια στην οικονομία. Εάν δεν θέλετε, αυτούς που δεν θέλετε να φορολογήσετε είναι οι κερδοσκόποι με το high frequency trading που μετακινούν δισεκατομμύρια και κάνουν την οικονομία μας απρόβλεπτη απρόβλεπτη και εις βάρος του καλού επιχειρηματία, του καλού επενδυτή που θέλει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Γι' αυτό η θέση σας δεν αρκεί και πρέπει να βρούμε τη δική μας φωνή. Κύριε Γκοζές, λυπούμε. Σας εκτιμώ κατά τα λοιπά, ως συνάδελφο, αλλά εδώ πέρα έχετε άδικο. Έχετε άδικο γιατί αποδυναμώνει τη θέση του Κοινοβουλίου που είχαμε από τη θέση συμπερέ. Αποδυναμώνει ε, τη θέση μας ο κύριος Γκοζές και όποιο συμφωνεί μαζί του θα φροντίσει η Κομισιόν να εξακολουθεί να κάνει αυτό το οποίο θέλει, δηλαδή να μην προτείνει τέτοιο φόρο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των θέσεων Γκοζές. Γι' αυτό είναι λάθος να τον ακολουθήσουμε αυτή τη φορά, αγαπητοί συνάδελφοι. Όποιο θέλει να δώσει φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρώπης, να ξανακοιτάξουμε ελπίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πιστεύουν πως κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, πρέπει αυτή τη φορά να ψηφίσει το εναλλακτικό ψήφισμα των σοσιαλδημοκρατών και τροπολογία 2 την οποία υπέγραψαν πάνω από 120 συνάδελφοι από όλες σημαντικές ε, κοινοβουλευτικές ομάδες. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ συνάδελφος Όλες Μη των ε, Φιλελευθέρων και Δημοκρατών έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ποδηματά για την έξοχη συνεργασία μας και πραγματικά πετύχαμε συμβιβασμό παρά τις διαφορές που είχαμε μεταξύ μας. Σήμερα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτό το συμβιβασμό επί το οποίου τοποθετήθηκε και η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Και το λέω και στον κύριο Μπούλμαν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτή η έκθεση να δημιουργήσει πραγματικά μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη όπως χρειάζονται και προγράμματα υποδομών ε, μέσω των ευρωμολόγων. Ε, των ευρωπαϊκών αυτών αξιογράφων που θα μπορούσαν να, θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα φόρο όσον αφορά τον άνθρακα στην ευρωπαϊκή αγορά για να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τα κάτι μέλη, κατά την άποψή μου, θα πρέπει έχουν υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν σημαντικά έργα υποδομών. Στη χώρα μου, στη Σουηδία, η Σουηδία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που σέβεται τους στόχου αυτούς και ο χρηματοδοτικός τομέα σίγουρα θα πρέπει να συμμετάσχει ε, στις δαπάνες. Ε, δημιούργησε ο τομέα αυτός την κρίση για άλλους Ευρωπαίους πολίτε στο κάτω-κάτω. Η λύση όμως δεν είναι ο φόρο των οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μου, κύριε Πρόεδρε. Τη δεκαετία του 80 εισήχθη ένα είδος φόρος αυτού του είδους ε, και πολλοί εκπρόσωποι του τομέα, ε, φορείς του χρηματοστικού τομέα, το έσκασαν και πήγαν στο Λονδίνο. Δεν θα πρέπει να επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο της Σουηδίας σε όλη την Ευρώπη. Δεν λέμε ότι οι διαστάσεις ίδιες, αλλά πολύ γρήγορα κινούνται αυτοί τα χρήματα. Υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, δεν πιστεύουμε ότι ο φόρος των οικονομικών συναλλαγών ε, μπορεί να αποτελέσει λύση. Σύμφωνα με την ομάδα ALDE, αυτό ο φόρο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορέσει να έχει θετικέ ε, συνέπειε. Η ομάδα μα, κύριε Πρόεδρε, λέει όχι στην τροπολογία 1 και 2. Αντίθετα, μπορεί να αποδεχτεί την τροπολογία 3 ε, του κυρίου Γκοζέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφοι. Κύριε συνάδελφοι, εκ μέρου των Πρασίνων, ο Φιλίπ Λαμπέρτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ γιατί μιλάμε για τους καινοτόμους πόρους ξαφνικά ε, έχουμε μπει στο παιχνίδι του φόρου, όχι. Ε, τα δημοσιονομικά πρέπει να ανακάμψουν ε, με βιώσιμο τρόπο. Χρειάζεται δαπάνη με υπεύθυνο τρόπο, αλλά χρειάζονται και έσοδα που είναι δίκαια και αποτελεσματικά και βιώσιμα. Και το γνωρίζετε, τα φορολογικά συστήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη σήμερα δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια. Οι κυβερνήσει δεν έχουν τα μέσα για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο τομέα, όπω είναι η διδασκαλία, η έρευνα, η κοινωνική συνοχή. Δεν έχουν του πόρου, δεν μπόρεσαν να, ε, δεν μπόρεσαν να καλύψουν τι ανισότητε στην Ευρώπη και συνεχίζεται η καταστροφή τη κοινωνική συνοχή και η καταστροφή του περιβάλλοντο. Τώρα είτε φορολογήσουμε το χρηματοδοτικό τομέα, είτε έχουμε σωστή συμβολή από τι μεγάλε επιχειρήσει, ή αν θέλουμε να έχουμε ένα φόρο για το κλίμα και την ενέργεια για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά και τη φοροδιαφυγή, και αν τα κάνουμε όλα αυτά, για να τα πετύχουμε αυτά, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να τα πετύχουμε για να έχουμε αποτελεσματικέ λύσει σε επίπεδο 100 μελών είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ακούσαμε επί, ε, πρέπει να βρούμε σωστή κοινή προσέγγιση. Ούτε και 10 χρόνια να περάσουν δεν μπορεί μόνη της μια χώρα μέλος να βρει τους αναγκαίους πόρους. Πρόκειται η σωστή οικονομική διαχείριση. Θα πρέπει στα κράτη-μέλη να πούμε τι να κόψετε τις δαπάνες και δένοντας το χέρι από πίσω των εσόδων από την άλλη παιδιά. Κόψτε τις δαπάνες και κόψτε και τα έσοδα. Πώ να πολεμήσει κανεί με ένα δεμένο χέρι και ένα κομμένο χέρι. Η έκθεση τη κυρία Ποδηματά ανοίγει διόδου που μπορούν να βρουν απαντήσει όσον αφορά το πρόβλημα τη φορολογία και ελπίζω να υιοθετήσει αυτή την έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα έχουμε τον κύριο Ιβο Στρέιτσεκ από του συντηρητικού και που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ. Ξέρετε πως ε, αυτή τη στιγμή επιτάπητος ε, έχουμε τον φάκελο αυτό που λέγεται καινοτόμος ε, χρηματοδότηση. Νομίζω πως μπορούμε να πράγματι να μιλήσουμε για την εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων και ξέρουμε εκ των προτέρων και ποιος θα τους πληρώσει. Οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να κατηγορούμε τις τράπεζες πως ε, προκάλεσαν ε, την κρίση γιατί γνωρίζουμε πως υπάρχουν οικονομικές ανισορροπίες ε, παγκοσμίω και ξέρουμε ποιος φταίει γι' αυτό. είναι δυστυχώς οι πολιτικές παρεμβάσεις και η υπερβολική ρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα. Δεν νομίζω πως μπορούμε εδώ πέρα να φορολογήσουμε τόσες πολλές συναλλαγές των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Και εξάλλου όταν εισάγονται νέοι φόροι το πιθανότερο είναι πως ο τομέας αυτός θα τροποποιήσει ανάλογα την συμπεριφορά του και θα μετατοπίσει την έδρα του κάπου αλλού και αυτό θα είναι εις βάρος μας. Και εάν ε, ε, γίνει αυτό θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι θα μείνουν εδώ πέρα, δηλαδή οι ε, πελάτες. Ειδικά λοιπόν σε χρόνους πάρα πολύ μεγάλων οικονομιών στον προϋπολογισμό δεν θα έπρεπε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προχωρούν σε τέτοιες πράξεις ειδικά όταν δεν ε, κάνουν περικοπές. Αντιθέτως μιλάνε για νέους φόρους. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν ε, να κλείσουν κάποιες από τις ε, πολυέξοδες αυτές αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να χρηματοδοτήσουμε κάποιο ευρωπαϊκό έργο. Επίσης κάτι ακόμα για τα ευρωομόλογα αν εγκριθούν θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά φαίνεται πως έτσι θα τις αποφύγουμε. Θα υπάρχει συνεχώς κάποιος ο οποίος θα πληρώνει και θα υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Εμείς λοιπόν είμαστε κατά. Ο κύριος Κλούτε έχει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η απέτηση για φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών δεν είναι κάτι το νέο. Εμείς που ήμασταν κατά της παγκοσμιοποίησης το ζητούσαμε. Βέβαια πριν από πέντε χρόνια δεν το πίστευε κανείς. Αλλά αυτή την εβδομάδα είναι στη μερίσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί με ένα φόρο ε, για το δεξίο του άνθρακα και τα ευρωμόλογα και αυτό το βρίσκω θετικό. Τα οικονομικά μέσα τα οποία προτείνει η κυρία Ποδηματά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να στηρίξουμε και βέβαια θα τα ε, υπερψηφίσουμε. Είναι μέσα τα οποία χρειαζόμαστε άμεσα, καθώς ε, μέχρι τώρα οι προπολογισμοί επικεντρώθηκαν μόνο στο να περικόπτουν τα έξοδα, όμως τα δημόσια έξοδα και η περικοπή τους πληρώνει φτωχούς εργαζόμενους και συνταξιούχους, αυτούς τους οποίους είναι εξαρτημένοι από το κοινωνικό κράτος και έχουμε παραβλέψει τελείως τα έσοδα τα οποία βεβαίως μπορούμε και αυτά να εκμεταλλευτούμε, αλλά θα πρέπει κυρίως να στραφούμε σε αυτούς οι οποίοι προκάλεσαν την κρίση. Για να υπάρξει λοιπόν εξυγίανση των προϋπολογισμών θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν τα έσοδα Βεβαίω, μην ξεχνάμε πω εδώ πέρα υπήρχε μια κρατικοποίηση ιδιωτικών χρεών, των χρεών των τραπεζών και υπήρχε η χρηματοδότηση τη ε, τραπεζική κρίση από τον δημόσιο τομέα. Οπότε δεν είναι το κράτο αυτό το οποίο έχει την ευθύνη για την οικονομική κρίση και απαιτείται πολιτικά να πληρώσει επιτέλου ο χρηματοοικονομικό τομέα. Με τον φόρο λοιπόν αυτόν επιτέλου αυτό ο οποίο προκάλεσε την κρίση δημοσίου χρέου ε, θα βοηθήσει και να πληρωθεί αυτή η κρίση. Αυτό είναι σημαντικό πολιτικό μήνυμα, εάν ε, εγκριθεί αυτή η έκθεση όπως έχει υποβληθεί. Αλλά και τα ευρωομόλογα θεωρούμε πως είναι ένα αξιόλογο και χρήσιμο μέσο, γιατί συνεισφέρουν περισσότερο από όλε τις κυρώσεις στη μείωση και τις συμβουλές στη μείωση των ε, χρεών. Επίσης, δεν είναι ε, από την άλλη αποδεκτό οι χώρες οι οποίες έχουν τα πλεονάσματα ε, να εκμεταλλεύονται την ε, όλη κατάσταση. Βεβαίω μπορούμε να ασκήσουμε κριτική και να πούμε πως είναι μία αναδιανεμητική ένωση, αλλά όποιος θέλει κοινωνική Ευρώπη θα πρέπει επί της αρχής τουλάχιστον να είναι υπέρ μιας ε, τέτοιας πολιτικής. Επίσης θέλω να πω στην Κομισιόν πως ελπίζω πως ε, επιτέλους θα υποβάλει προτάσεις ε, για έναν τέτοιο φόρο, τις οποίες έχουμε ζητήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάρατς ε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η θεωρία για ένα φόρο Tobin κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια έναν παγκόσμιο φόρο για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, αλλά δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Αυτό το οποίο προτείνεται σήμερα εδώ και επειδή ε, είναι απελπισμένη για χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται και ίδιους πόρους. Αυτό το οποίο προτείνεται εδώ λοιπόν είναι ουσιαστικά ε, μια δυνατότητα να ε, ταράξουμε τα νερά στο χρηματοπιστωτικό δομή που δεν είναι καθόλου δημοφιλής και νομίζουμε ότι όλα αυτά θα μας φέρουν έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπούμε πολύ όμως ζούμε σε παγκόσμια οικονομία κυρίες και κύριοι και αν καταστούμε μη ανταγωνιστικοί μέσω φορολογικών ρυθμίσεων πολύ απλά ο κόσμος θα μετακινηθεί και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 24 ώρες. Άρα αν κάνουμε κάτι τέτοιο ουσιαστικά είναι οικονομικά καμικάζι η μεγαλύτερο τομέα, ε, ο χρηματοπιστωτικό ε, στον κόσμο είναι στο Λονδίνο. Και αν δεν ε, τα ήξερα καλύτερα, θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία να σταματήσουμε του Αγγλοσάξονε να κάνουν τι δουλειέ του. Το 2010, λόγω τη οδηγία AIMF, ένα από τα τέσσερα hedge funds έφυγε όμω από το ΣΥΤ του Λονδίνου. Και αν συνεχίσουμε την ίδια κατεύθυνση, η Βρετανία θα έχει χάσει τη μεγαλύτερη βιομηχανία, το μεγαλύτερο κλάδο τη. Και κάποια στιγμή το ΣΥΤ χρηματοπιστωτικές αγορές θα στραφούν, θα εξεγερθούν κατά της συμμετοχής της χώρας τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το ψηφίσουμε λοιπόν, ίσως αυτό θα ήταν εν τέλει καλό για, το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν θέλουμε να είμαστε μέλος αυτού του πειράματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Μάρτιν Έρενχάουζερ. Κύριε Φάρατζ, δεν έχετε δίκιο. Εγώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εδώ πέρα να αποδείξει να αξία της. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω μπορεί αύριο στην ψηφοφορία, εάν υπερψηφίσουμε όλοι, να γίνει ένα νέο σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτού του φόρου και μπορεί να δώσει και η πολιτική το μήνυμα ότι θα σπάσει τις αλυσίδες σκλαβιάς από τον οικονομικό τομέα. Όμως αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει μόνο μια αφορμή προς τον οικονομικό τομέα για να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις με αξία στην πραγματική οικονομία. Όχι, πρέπει να φύγει και το φορολογικό βάρος από τον εργαζόμενο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θάρρος, θάρρος εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικά όταν ορίζουμε το ποσοστό όταν μιλάμε για 0,03 ή 0,05% δεν επαρκεί. Πρέπει να θέσουμε έναν στόχο τουλάχιστον ή μέχρι το 0,5% και αν ναι ε, τότε εγώ οπωσδήποτε θα ψηφίσω και την ε, τροπολογία. Δύο ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε, για τις δηλώσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάμε για καινοτόμο χρηματοδότηση, αλλά επειδή έχουν ήδη ακουστεί μερικά πράγματα, καινοτομία δεν είναι μόνο να εφευρίσκουμε νέους φόρους ή παλαιά πράγματα όπως ε, το κρατικό χρέος να τα ονομάζουμε με άλλο όνομα. Αλλά θα ήθελα τώρα να περάσω στην ουσία. Η ουσία δεν είναι τα ευρωομόλογα. Κάτι ε, είμαστε, εξάλλου κατά και των ευρωμολόγων τη Τσέσου. Πρέπει να βγάλουμε τα συμπεράσματα από την οικονομική κρίση και τα συμπεράσματα πολύ απλά είναι πω η κερδοσκοπία πρέπει και αυτή να φορολογηθεί. Και αυτό σημαίνει, θέλω να το πω σαφώ εάν δεν γίνεται παγκοσμίω ή σε επίπεδο G20, να το κάνουμε εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει, πιστεύω, καμία εναλλακτική. Γι' αυτό Κύριε Μπούλμαν, μην χειροκροτείτε μόνο τώρα, αλλά ελπίζω αύριο να έχουμε ισχυρή πλευσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Κομισιόν ω σύμμαχο κατά των κρατών μελών, ειδικά κατά των κρατών μελών που ακούσαμε τώρα να μιλάνε τόσο δυνατά και σκέφτονται τι θα γίνει με το City του Λονδίνου. Θα σα πω μόνο το εξή, κύριε Φάρατζ. Δείτε τα νούμερα των ανέργων, την οικονομική καταστροφή της χώρας σας, που επικεντρώθηκε μόνο σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Αν φτιάχνετε και κάνα αμάξι όπως εμείς στη Βαβαρία και στη Γερμανία θα πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό απαιτείται να εισαχθεί τώρα αυτός ο φόρος, να τον απαιτήσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι αυτό θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Λονάρντο Ντομένιτς έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση της κυρίας Ποδηματά εμπεριέχει έχει πολλές σημαντικές πτυχές που δεν περιορίζονται μόνο στο θέμα της φορολογήσεως των οικονομικών συναλλαγών. Είναι πλούσια έκθεση, είναι πλούσια σε προτάσεις και σε ανάλυση και ελπίζω να υποστηριχθεί ευρέως από το Κοινοβούλιο είναι ενδεχομένω η βάση για μια πραγματική νέα φορολογική πολιτική, ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική που τη χρειαζόμαστε. Αν μιλάμε για φορολογική εναρμόνιση και σε αυτή την έκθεση υπάρχουν προτάσεις που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση μιας φορολογικής εναρμονίσεως που δίνει νέα ισχύ ε, και νέο πρόσωπο στην Ευρώπη. Είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση η συζήτηση επικεντρώνεται πάνω απ' όλα στο φόρο επί των χρηματοσυντικών συναλλαγών που θα εφαρμοστεί σαν ένα πρώτο στάδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτή είναι η στιγμή θαραλέων επιλογών που θα πρέπει να εφαρμοστούν με ισορροπημένο τρόπο, αλλά θα πρέπει να ανοίξουν ένα δρόμο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει την αρμοδιότητα να δείξει ένα δρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτό το Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα καθήκον να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα. Να πω ένα πράγμα στον κύριο Σμιτ τον οποίον σέβομαι πολύ. Σέβομαι και ε, το ξεκάθαρο μυαλό του και την ευφία του. Πρέπει να προσέχουμε τι επιχειρήματα χρησιμοποιούμε σήμερα. Αν πούμε σήμερα ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το φορο των χρηματοστικών συναλλαγών, διότι υπάρχουν οι φορολογικοί παράδεισοι, θα δώσουμε την εντύπωση στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε αφοπλισμένοι τη στιγμή που πολλά από αυτά τα χρηματοστικά ιδρύματα ξανάρχισαν να βγάζουν κέρδη. Και αυτή δεν είναι μία η πρόταση των σοσιαλιστών στη χώρα μου, στην Ιταλία. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε και από πολλές, πολλές αυτόνομες ενώσεις και υποστηρίχθηκε και από το καθολικό και δημοκρατικό κίνημα υπέρ της ανάπτυξης και ισορροπημένης εξέλιξης και ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σιλβί Γκουλάρ έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να χαιρετήσω το έργο της συναδέλφου μας της κυρίας Ποδηματά που πράγματι επετέθη επί πολλών ευαισθητών θεμάτων. Δεν θα αναφερθώ στα ευρωμόλογα που αναφέρω στην έκθεσή μου για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Θα ήθελα να θέσω τρία ζητήματα όσον αφορά το φόρο των χρηματοδοτικών συναλλαγών. Το πρώτο θέμα, χρειαζόμαστε νέα έσοδα και έχουμε το δικαίωμα σε αυτό το κοινοβούλιο να μιλάμε από καιρού καιρών όσον αφορά την πτυχή αυτή των εσόδων. Η απάντησή μου είναι ναι, υπάρχουν ταμπού στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνουμε συνολικό προβληματισμό για διέξοδο από την κρίση αν δεν είμαστε σε αν δεν είμαστε ικανοί, και εδώ χαιρετίζω το έργο που έκανε και ο Επίτροπο ο κ. Σεμέτα όσον αφορά του άλλου φόρου, για να αντιμετωπίσουμε, λέγω, αυτό το θέμα χωρί ταμπού. Δεύτερον, χρειαζόμαστε το φόρο όσον αφορά τι χρηματοστικέ συναλλαγέ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση και θα σπεραπέμπω σε μια δουλειά που πρόσφατα έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε διαβουλ... μετά από διαβουλεύσεις που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη όσον αφορά το MIFID όλα τα κείμενα που αφορούν το high frequency trading δηλαδή τις συναλλαγές τις πολύ γρήγορες που κάνουν οι υπολογιστές εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πρόσφατες επικίνδυνες εξελίξεις και συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος Φέρμπερ όσον αφορά το ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δράσεων της αγοράς που επιτρέπουν την ρευστότητα και δράσεων πιο κερδοσκοπικών και ενδεχομένως επιβλαβών. Τρίτο σημείο, και αυτό το τελευταίο σημείο μου, χρειαζόμαστε παγκόσμιους κανόνες ή ευρωπαϊκούς. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω τι σημαίνει παγκόσμιους κανόνες. Θα περιμένουμε και τελευταία δικτατορία του κόσμου να συμφωνήσει για να αποφασίσουμε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρυβόμαστε πίσω από την παγκοσμιοποίηση για να μην επομιστούμε τις ευθύνες μας. Νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά παράλογο κάτι τέτοιο και από ό,τι φαίνεται χρειαζόμαστε να λάβουμε υπόψη τους κινδύνους της ε, μεταγκατάστασης και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Και από την άλλη πλευρά το Κοινοβούλιο δεν αποφάσισε όσον αφορά την ε, απειλή αυτή. Θα πρέπει να μια απόφαση. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σβέν Γκίγκολντ έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Er- ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ την κυρία Ποδηματά. Δεν ήταν εύκολο αυτό το οποίο έκανε. Τις τελευταίε εβδομάδες παρατηρήσαμε τα email που λάβαμε, την έντονη συζήτηση και εντό κάποιων ομάδων, πως αυτό το θέμα απασχολεί και πάρα πολλού πολίτε και παρατηρούν πώς τοποθετούνται οι πολιτικοί στο κοινοβούλιο αυτό για το θέμα. Ο φόρος αυτός είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών που είχε ξεκινήσει από την ε, πρόταση Τόμπιν, φόρου Τόμπιν και άρα είναι αποφασιστικό το πώς θα κινηθεί το Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά λοιπόν το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να είναι παγκόσμιος ο φόρος και δεν υπάρχει αντίπαλος στο παγκόσμιο επίπεδο. Το επόμενο ερώτημα είναι θα έπρεπε να εισαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτός ο φόρος και εκεί πέρα πρέπει να πούμε πως πολλοί από τους αντίπαλους ε, κρύβονται πίσω από το επιχείρημα αυτό και ακριβώς θα πρέπει να το απορρίψουμε αυτό. Γιατί Ήδη και σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν επιτυχείς φόροι συναλλαγών οι οποίοι λειτουργούν για μεμονωμένες αγορές. Δηλαδή ακόμα και αν ο κύριος Σεμέτα επεξεργάζεται την ε, μελέτη επιπτώσεων δεν απαντάει αυτό στο ερώτημα εάν μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιος φόρος, αλλά σε ποιες μεμονωμένες αγορές μπορεί να λειτουργήσει, σε ποιος ε, μπορεί να λειτουργήσει ε, πανευρωπαϊκά και σε ποιες μόνο παγκοσμίω. Οπότε, για όλους όσους θέλουν, θέλουν να φορολογήσουν τις συναλλαγές, δεν υπάρχει λόγος αύριο να καταψηφίσουν την διατύπωση ε, των 120 βουλευτών. Οπότε σας ζητώ κύριε Σέμετα τελειώστε την μελέτη σας αυτή, παρατηρήστε πόσο μεγάλη είναι η υποφορολόγηση αυτού του τομέα και αύριο αγαπητοί συνάδελφοι ας στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για έναν τέτοιο φόρο. Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος κατά. Κύριε Χίλτα Φιγκερέδη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένας φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι καιρό που συζητείται και συζητείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά να πάψουν να ισχύουν αυτή η φορολογική παράδειση και η κερδοσκοπία εδώ και ε, καιρό, καιρό. γίνεται λόγος για αποτελεσματικό έλεγχο και ρύθμιση των κεφαλαίων αγορών για να μην υπάρχει κερδοσκοπία μεταξύ προϊόντων πρώτων υλών, ακινήτων, συντάξεων, ασφαλίσεων κτλ. Ε, μιλάμε για ένα ολόκληρο πλωστάσιο παραγόγων επίσης και μιλάμε και για τα ε, κυρίαρχα δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάνει τις προτάσεις της αλλά νομίζουμε ότι οι χρηματοπιστωτικές απώλειες στην Ευρώπη είναι γύρω στα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα δημόσια ελλείμματα χωρίς καν να αυξήσουμε τους φόρους. Οι εκτιμήσεις που γίνονται σήμερα για τα έσοδα τα οποία θα μπορούσαν να προέλθουν από έναν φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα μας έδιναν πάνω από 2 δις ευρώ ετησίως. και 650 ε, εκατομμύρια ε, δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί καθυστερούμε, γιατί καθυστερούμε ένα τέτοιο φόρο λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει αυτό το πρόσχημα, θέλετε, να κάνουμε νέες μελέτες, αναλύσεις. Εγώ νομίζω όμως ότι